τη ψαλίδα του εσόδου ε, ανοίγει. Χρειάζεται δηλαδή περισσότερα έσοδα γυναίκες, θα πρέπει να συμμετέχουν και οι πατέρες τους. Ευχαριστώ λέει πρόεδρος, ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση και η έκθεση κυρία Στελάχ θα ψηφιστεί στις 12.30 την Δετάρτη και η έκθεση κυρία Τόμψεν ήδη αύριο στις 12.30. Λοιπόν, Αγαπητοί συνάδελφοι, το επόμενο σημείο τη σημερινή είναι η κοινή συζήτηση για τη συμφωνία πλαίσια μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλου και τη Επιτροπή. Πρόκειται για δύο εκθέσει του κ. Ράγκελ. Καταρχήν, η αθεώρηση τη συμφωνία πλαίσια για τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή και η προσαρμογή του κανονισμού του Κοινοβουλίου στην αναφερμένη συμφωνία πλαίσιο για τη σχέση μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη Επιτροπή. Ο εισηγητής έχει το λόγο. Τέσσερα λεπτά κύριε Ράγγελ, παρακαλώ. <coughs> Äh, äh, κύριε Πρόεδρε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι όσον αφορά τα δύο αυτά σημεία που συζητούμε, να πω εκ μέρους της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων ότι ο κ. Λένε, ο κ. Βόμποντα, η κυρία Ροτ Μπέρεν, η Νταϊάννα Βάλλη και η κυρία Χάρμ κάνανε έξοχη δουλειά. Ε, αποτελούσαν την ομάδα του Κοινοβουλίου που διαπραγματεύτηκε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη συγκεκριμένη συμφωνία. Θα ήθελα να τονίσω επίση ότι επεκράτησε πνεύμα ανοιχτό και επικοδομητικό από πλευρά του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από τον Επίτροπο Σεφκοβίτς και το προσωπικό του πετύχαμε αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Πετύχαμε μια ιστορική συμφωνία που είναι η πρώτη συμφωνία πλαίσιο μετά από την θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας. Η πρώτη συμφωνία πλαίσιο που βασίζεται άμεσα σε συγκεκριμένη νομική βάση που περιγράφεται στην συνθήκη. Το άρθρο 109, πιο συγκεκριμένα, που αφορά τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Νομίζω, λοιπόν, ότι οι σχέσεις μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, έχουν γίνει αρκετά στενές. Κατελήξαμε σε ένα συμβιβασμό, πετύχαμε μια ισορροπία όσον αφορά τις θέσεις των ε, θεσμικών οργάνων και το ρόλο που διαδραματίζουν στα πλαίσια της ε, νέας συνθήκης. Η διαπραγματευτική ομάδα ε, εργάστηκε στα πλαίσια θετικού πνεύματος και στη συμφωνία πλαίσιο καταφέραμε να πετύχουμε την αύξηση των εξουσιών μας ε, δυνάμει της συνθήκης της Αβώνας όσον αφορά και την ε, νομοθετική διαδικασία και την οργάνωση των εργασιών. Αυτά είναι απλώς δύο παραδείγματα. Και όσον αφορά την τοποθέτησή μας αφορά το πρόγραμμα εργασιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και την χρήση των, της ήπιας νομοθεσίας, όπου εκεί οι νομοθετικές αρμοδιότητες του Κοινοβουλίου ε, έχουν επιρροή. Δεύτερο σημαντικό σημείο είναι η ενίσχυση των εξουσιών του Κοινοβουλίου για έλεγχο. Καθορίζοντας τους κανόνες για τον Πρόεδρο και τα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τις εμφανίσεις του στο Κοινοβούλιο και τη δυνατότητα να ε, αφαιρεθεί εξουσία από έναν επίτροπο, να διωχθεί από τη θέση του και τη συμμόρφωση με τις διεθνείς συνθήκες και τις συνομιλίες. Σε όλες αυτές τις πτυχές το Κοινοβούλιο είχε εξουσία βάσει της θήξης της αγώνας ε, η πρόσβαση στις πληροφορίες έχει μεγάλη σημασία επίσης και η πρόσβαση σε απόρριτες εμπιστευτικές πληροφορίες. Πέραν αυτού και ανταλλαγή πληροφοριών και ανταλλαγή απόψεων καλύπτονται ανταλλαγές μεταξύ εκπροσώπων του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Γνωρίζουν παραδείγματι ότι σήμερα είναι δυνατόν ο Επίτροπος, υπεύθυνο για συνταγματικά ζητήματα, να παρίσταται στις συνεδριάσεις της διασκέψεως των Προέδρων όταν συζητούνται τέτοια θέματα και υπάρχει και διάλογος μεταξύ της διασκέψεως των Προέδρων των Προέδρων των Επιτροπών και παρουσίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Κοινοβούλιο, στις εργασίες του Κοινοβούλιο. Έχει ενισχυθεί λοιπόν αυτή η σχέση χάρη στην ώρα των ερωτήσεων, που δεν αφορά μόνο τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υποβολή ερωτήσεων, αλλά και τα μέλη τη Ευρωπαϊκή Επιτροπής, τους Επιτρόπους. Σε πλήρη σεβασμό τη συνθήκη τη Αβώνας, που εμπεριέχει διατάξει για την ισορροπία δυνάμεων μεταξύ των θεσμικών οργάνων, καταλήξαμε σε μια συμφωνία που ξεκαθαρίζει την κατάσταση και η οποία συμφωνία θα εξασφαλίζει ότι η συνθήκη της Λισαβόνας πραγματικά θα τίθεται σε ισχύ με ζωντανό τρόπο. Ευχαριστώ. Επίτροπο Σεύκοβιτ, έχει τώρα το λόγο. Σα ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Εξότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Είναι μεγάλη χαρά μου να μπορέσω να συμμετέχω στη συζήτησή σα για την αναθεώρηση τη Συμφωνία Πλαισίου για τη σχέση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων και χαίρομαι που το ψήφισμα που θα υιοθετήσετε μεθαύριο ε, συστήνει στο Κοινοβούλιο να υποστηρίξει την ε, πρόταση αυτή. Μετά την θέση ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα, ε, εγώ θα ευχαριστήσω τον κύριο Λέμε, Λένε και την, θέση εργασία, την ομάδα εργασία, την κυρία Νταϊάννα Βόλη, την κυρία Ντάγμαρ Πέρεν, Ρεμπέκα Χάρμ, Χάνε Βόμποντα και βέβαια τον εισηγητή Παόλο Ραντζέλ γιατί συνεργάστηκαν πάρα πολύ καλό και έντονα. Οι συζήτησει μας ήταν πάρα πολύ φιλικές αλλά και επικοδομητικές. Είναι προφανές ότι η αύξηση των αρμοδίτων του Κοινοβουλίου μετά τη νέα συνθήκη έχουν επιπτώσεις στις σχέσεις εργασίας μεταξύ των θεσμικών οργανών. Αυτό ανεκαθρίζεται και από το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 9 η Φεβρουαρίου τρέχοντας έτος και την κατόπιν δήλωση του Προέδρου Παρόζο την ίδια μέρα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό με τον θεωμένη συμφωνία πλαίσιο να έχουν τα θεσμικά μας όργανα τώρα μία ε, επίσημη βάση για τις αμοιβαίες σχέσεις και να αρχίζουν να εφαρμόζονται όλα τα στοιχεία της συμφωνίας καθημερινά. Αυτή η ανθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο βασίζεται στην ισχύουσα συμφωνία πλαίσιο του 2005 που από ό,τι είδαμε ήταν πάρα πολύ ε, επιτυχές μέσο για την ε, βάσιση των σχέσεων μεταξύ των δύο οργάνων. Πάνω σε αυτόν, σε αυτή τη θετική εμπειρία βασίζαμε τις διαπραγματεύσεις μας για την ανθεώρηση του σχεδίου πλαισίου το Μάρτιο και θα είμαστε όλοι ικανοποιημένοι νομίζω με το αποτέλεσμα. Όπως και ο εισηγητής σας ο κ. Ραντζέλ, έτσι και εγώ θεωρώ ότι η αναθεώρηση αυτή είναι μια σημαντική ε, ένα σημαντικό επίτευγμα για τη σχέση μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων λάβαμε ω υπόψη τη νέα αρμοδιότητα του Κοινοβουλίου μετά τη ισχύ τη συνθήκη του Λισαβόνα. Έτσι προωθείται η καλύτερη σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής, Ένωσης, Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Κοινοβουλίου. Πού υπάρχει σημαντική πρόδρος. Η συμφωνία καθορίζει χρονοδιάγραμμα και κανόνες για την ενδυνάμωση των σχέσεών μας που θα επιτρέπουν στο Κοινοβούλιο να συμβάλλει σημαντικά όταν η Κομισιόν προετοιμάζει το πρόγραμμα εργασία τη, Καθορίζει συγκεκριμένου και λεπτομερεί κανόνε. Το θα κάνει η Κομισιόν για τις διαπραγματεύσει και την ολοκλήρωση των διεθνών συμφωνιών. Αναφέρεται σε κανόνες για την χορήγηση ε, προστατευόμενων πληροφοριών, απορρίτων πληροφοριών προς το Κοινοβούλιο, πώς θα ενημερώσει παραδείγματος το Κοινοβούλιο για την συνέχιση διεθνών διαπραγματεύσεων. Αναφέρεται επίσης πώς θα δοθούν οι πληροφορίες στο Κοινοβούλιο για την ενημέρωση που λαμβάνει η χώρα στην Επιτροπή από ερυπηρευνόμονες. Θα εξακολουθούμε να έχουμε, να έχουμε τη δυνατότητα να σας προσφέρουμε εδώ την παρουσία των επιτρόπων. Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες παρατηρήσεις όσον αφορά την προετοιμασία του προγράμματος εργασίας 2011 για την Κομισιόν. Στη διασ... Ο κ. Παρόζο έκανε μια παρουσίαση. Εγώ πήγα στη διάστηση του Προέδρου και έκανε μια σχετική παρουσίαση. Το... 7 Οκτωβρίου συναντήθηκε η διάσκεψη του Προέδρου με το συλλογικό όργανο της Κομισιόν. Αυτό θα ξαναγίνει την επόμενη εβδομάδα. Αυτό καταδεικνύει πόσο σημαντική είναι αυτή η συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και νομίζω ότι πετυχαίνουμε έτσι τα σωστά μέσα στην συμφωνία πλαίσιο. Ξέρουμε μέρη, όπως ξέρετε, οι διαπραγματεύσεις για την αναθεώρηση της ε, συμφωνίας αυτής ήταν μακρές και απαιτούσαν σημαντικές προσπάθειες και από τις δύο πλευρές για να έχουμε ένα κείμενο που να λαμβάνει υπόψη όλων τις ανησυχίες. Ξέραμε επίση ότι για πολλέ από τι σχέσει μα, παραδείγματο χάνει το πρόγραμμα της ε, Ένωσης που εισάγει η συνθήκη του Πισταβόνου θα πρέπει να παίξει ρόλο και το Συμβούλιο. Το Συμβούλιο δεν θα είναι τμήμα των διαπραγματεύσεων για την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο. Γι' αυτό φροντίσαμε να μην προδικάσουμε θέματα που πρέπει να συμφωνηθούν στο Συμβούλιο. Γι' αυτό οι διαπραγματευτές και από τις δύο πλευρές καταβάλουν σημαντικές προσπάθειες για να πετύχουν την, να διατηρηθεί η ισορροπία μεταξύ των θεσμικών οργάνων όπως καθορίζεται και από τη συνθήκη. Αυτό αναφέρεται συνεχώς στη συμφωνία. Επίσης η ε, Κομισιόν θεωρεί ότι το κείμενο που επετεύχθη μετά από δύσκολες εν μέρη διαπραγματεύσεις σέβεται απόλυτο τα δικαιώματα και αρμοδιότητες των θεσμικών οργάνων και μπορεί πραγματικά να ελεγχθεί σε όλες τις λεπτομέρειες. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι η Συμφωνία Πλώσιο λένε πολύ πάει πολύ μακριά και ότι η νομική πίεση δεν μπορεί να αποκλειστεί. Γι' αυτό η Κομισιόν σημειώνει ότι η πρόταση ψηφίσματος για την υιοθέτηση της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαίσιο θα καθορίσει επίσημα την κοινοβουλευτική ερμηνεία του κειμένου αυτού. Πολλές φορές αυτές οι συμφωνίες ξεπερνάνε το συμφωνημένο κείμενο μετά από πολλέ πληροφορίε, παραδείγματο χάρη όσον αφορά την ενημέρωση του Κοινοβουλίου για τι διαπραγματεύσει για την Εθνική Συμφωνία, καθώ επίση τη συμμετοχή ευρωβουλευτών σαν παρατηρητέ στι διεθνέ αυτέ διακέψει. Στην Επιτροπή η Κομισιόν είπε ότι αυτές οι προσπάθειες έχουν σαν στόχο να σημειώσουν απλώς τις αρχικούς ε, ε, στόχους του Κοινοβουλίου. Για να μην υπάρχουν αφιβολίες, η Κομισιόν έτσι δέχεται την ερμηνεία του Κοινοβουλίου για το κείμενο αυτό. Αξιότιμοι βουλευτέ, η Κομισιόν παραμένει αυστερά προσκολλημένη σε όλε τι δεσμεύσει που αναλυφθούν μέσω τη συμφωνία και σκοπεύει να εφαρμόσει τη συμφωνία αυτή βάσει του συμφωνημένου κειμένου. Θα ήθελα να είναι απόλυτα σαφές ότι η Κομισιόν δεν θα δεσμευτεί από μονομερείς ερμηνείες αυτού της συμφωνίας πλαίσιο. Το έγγραφο όπως έχει ε, τύχει αντικείμενο διαπραγματευτής πιστεύουμε ότι θα πρέπει να διασφαλίσει τα ε, δικαιώματα και συμφέροντα όλων. Θα πρέπει να σας πούμε ότι θα ελπίζουμε να υπάρχει στενή συνεργασία μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων. Προσβλέπω στην υπογραφή της συμφωνίας και την επιτυχή της εφαρμογή κατόπιν. Ευχαριστώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Σεφκοβιτ. Περνάμε τώρα στου ομιλητέ εκνόματο των πολιτικών ομάδων. Για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματο, ο κύριο Μέντε Τιβίκο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, εδώ και 18 χρόνια που ήταν συμβουλευτικό ο χαρακτήρα του, δεν είχε εξουσίε όταν ξεκίνησε και αυτή η διαδικασία αυτά τα 18 χρόνια έχουμε δει πώ το Κοινοβούλιο από συμβουλευτικό απλά έγινε συνομοθέτη. Όπω έλεγε και ο Φρανθίσκο Λούκα Πύρε, ε, ο φίλο μα, ε, ότι πλέον έχει και νομοθετικό ρόλο το Κοινοβούλιο. Αυτό το οποίο θα εγκρίνουμε την Τετάρτη λοιπόν ουσιαστικά είναι το αποκορύφωμα διαπραγματεύσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Συμφωνία Πλαίσιο. Και θα σας εμπιστευτώ το εξή. Όταν λέω στην οικογένειά μου ότι πάω στο Στρασβούργο και ότι του είπα συγκεκριμένα τώρα ότι θα έρθω για να μιλήσω για τη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Επιτροπή και Κοινοβουλίου, Χρειάστηκε να πω πάρα πολλά πράγματα να εξηγήσω γιατί σε επίπεδο εθνικών κοινοβουλίων αυτό δεν είναι κατανοητό. Γιατί πρέπει να υπάρξει συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπή για να εφαρμοστούν στην πράξη οι διατάξει των συνθήκων. Κι όμω πρέπει να γίνει και αυτό πρέπει να γίνει για έναν πολύ στοιχειώδη λόγο που τον είπε και ο Πάλο Ρανζέλ και, ως, ε, και ο Επίτροπο. Θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί. Ο στόχο, ο βασικό ε, τη ε, συμφωνία πλαισίου είναι εκ των προτέρων να επιλύσει και να καταργήσει εμπόδια τα οποία στο πλαίσιο τη και του κοινοβουλευτικού ελέγχου αλλά και των ε, κωδίκων συμπεριφορά θα μπορούσαν ε, να προκύψουν στην πράξη. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πρόκειται για ένα πολύ καλό μείγμα ευρωπαϊκής δημοκρατίας, ε, μιας συνενετικής δημοκρατίας που δεν βασίζεται σε συγκρούσεις όπως αυτές και αντιπαραθέσεις όπως αυτές που βλέπουμε στις χώρες μας. Και το ΕΦΙΕΣ, το έξυπνο, είναι ακριβώς να καταλήξουμε σε λύσεις για τα προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν. Αυτή λοιπόν η συμφωνία πλαίσιο για αυτούς τους λόγους είναι ένα μέσο που θα μας ε, ε, αποτρέψει να έχουμε προβλήματα στο μέλλον και που θα βοηθήσει την εφαρμογή των συνθήκων. Και δι έχουμε νέα συνθήκη, την συνθήκη της αγώνας εξού και έπρεπε να αναπτύξουμε αυτή τη ε, συμφωνία. Θέλω να ευχαριστήσω τον Ρανζέλ και την ομάδα του αλλά και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή γιατί φτάσαμε σε μια πολύ λογική συμφωνία. Διαβάζοντας αυτά που λέει η συμφωνία Εκπλήσεται κανείς ακούγοντας τις φωνές σε κάποια εθνικά κοινοβούλια που λένε ότι έτσι τίθενται σε κίνδυνο οι εξουσίες του Συμβουλίου. Μα οι εξουσίες του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο είναι ο άλλος συνομοθέτης. Ε, εμείς, αν ε, θέλουμε να συνομοθετούμε και τα κάνουμε πολύ καλά, συνεργαζόμαστε πολύ καλά με το ε, Συμβούλιο Υπουργών. Κοιτάξτε, δεν προσπαθούμε να αποκομίσουμε κάποιο μικρό όφελος, μικρό πλονέκτημα για το Κοινοβούλιο. Εμείς θέλουμε να είμαστε αποτελεσματικοί και εσείς πραγματικά κύριε Επίτροπε πιάσατε τον τάβρο από τα κέρατα όπως λέμε και στη χώρα μου που ασχολούμαστε και πολύ με τις σταυρομαχίες ό,τι αφορά ιδίως τα άθρα 6 και 7. Αυτό ακριβώς έτσι ερμηνεύει τα πράγματα και το κοινοβούλιο σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συνθήκες. Δεν υπάρχει κάτι περίεργο εδώ. Περί μας πρόκειται, θέλει το Κοινοβούλιο να ενημερώνεται και να συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις μέσω της Επιτροπής. Τίποτα περισσότερο. Να ξέρουμε τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλω λοιπόν να συγχαρώ και τα δύο θεσμικά όργανα και νομίζω, όπως θα έλεγαν και στο Λευκό Οίκο, είναι το, ε, η αρχή μιας ε, ωραίας νέας φιλίας. Ευχαριστώ. Τώρα θα ακούσουμε από, για, από τους σοσιαλιστές ε, τον κύριο Ατόντο. Για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε, θέλω και εγώ να συμφωνήσω με τους μέχρι τώρα προλαλήσαντε στη συζήτηση αυτή των τεχνικών δυσκολιών που ενδεχομένω έχει αυτή η συμφωνία, νομίζω ότι μιλάμε για κάτι σημαντικό. Για κάτι που θα πρέπει να το συνεξετάσουμε με τη μεταρρύθμιση να αναθεώρηση του κανονισμού πριν από κάποιους μήνες μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκη της Λισαβόνας. Μαζί λοιπόν αυτά τα δύο εργαλεία είναι δύο ουσιώδη στοιχεία της νέας δημοκρατικής αρχιτεκτονικής. Ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και νομίζω ότι ο νέο ρόλο αυτό που αναλαμβάνει με τη συνθήκη τη Λισαβόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γίνεται δηλαδή ένα νομοθετικό σώμα. Και με τι δύο συμφωνίε, τη μεταρρύθμιση του κανονισμού ε, και με τη συμφωνία πλαίσιο, το Κοινοβούλιο αποκτά ένα θεμέλιο, μία βάση, αν θέλετε, ε, λογική ε, για τη λειτουργία του. Και όπω υπόθηκε, είναι σημαντικό το Κοινοβούλιο από εδώ και πέρα ότι έχει τη λειτουργία και να διαλέγεται και να συμφωνεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο του νέου ευρωπαϊκού νόμου. Και για να γίνει αυτό χρειάζεται και ο νέο κανονισμό και η συμφωνία αυτή πλαίσια, η οποία καθορίζει όλα τα στοιχεία τα οποία διαμορφώνουν τι σχέσει μεταξύ των θεσμικών οργάνων. Γι' αυτό θέλω να τονίσω μεταξύ άλλων ε, την ε, εξουσία αυτή του κοινοβουλευτικού ελέγχου επί τη Επιτροπή. Κύριε Σεύκοβιτ, νομίζω ότι θα έπρεπε τελικά να εξετάσουμε το ενδεχόμενο κάποιων μηχανισμών παρουσίας της Επιτροπής ε, στο Κοινοβούλιο, όπως ε, προβλέπεται και στη Συμφωνία Πλαίσιο. Παρουσία όλων των Επιτρόπων, για παράδειγμα, για να απαντούν απευθείας στις ερωτήσεις μας, ώστε να υπάρχει μια άμεση ανταπόκριση στο πλαίσιο του πολιτικού μας ρόλου. Και σε ό,τι αφορά την ερμηνεία που κάνατε για τις παραγράφου 7 και 8, εγώ ήθελα να πω ότι την κατανοώ. Την κατανοώ την ερμηνεία αυτή, γιατί πράγματι δεν θα πρέπει να είναι μέρο, αυστηρά μέρο των διαπραγματεύσεων το Κοινοβούλιο. Πρέπει να καταλάβετε όμω ότι και εμεί ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουμε εκφράσει μια επιθυμία, μια θέση αρχή ω Κοινοβούλιο και στο μέλλον έχουμε εκφράσει το πώ θέλουμε να σχετίζεται και να συμμετέχει στι διεθνεί διαπραγματεύσει το Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ. Για τους φιλελευθέρους έχει το λόγο για δύο λεπτά ο κύριος Άντριου Ντάφ. Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή και ενδιαφέρον τον Επίτροπο Σεύκοβιτς. Φαίνεται ότι ενδιαφερόταν περισσότερο στο να καθησυχάσει το Συμβούλιο από ότι να επιτεθεί κατά της θέσης του Κοινοβουλίου με σοβαρότητα. Αυτό είναι σωστό, κατά την απόψή μου. Διότι αν το Συμβούλιο που βλέπω ότι δεν εκπροσωπείται, απουσιάζει απόψε, Εάν το Συμβούλιο, λέγω, ενδιαφερόταν σοβαρά να παίξει το ρόλο του και να γίνει μέρος της Συμφωνίας Πλαισίου, τότε το Συμβούλιο θα μπορούσε να το είχε κάνει. Σαν Κοινοβούλιο γνωρίζουμε ότι ενώ εφαρμόζουμε τις συνθήκες της Ζαβώνας θα πρέπει να ασκήσουμε τις νέες μας εξουσίες διακριτικά και υπεύθυνα. Επίσης, έχουμε δεσμευτεί στο να ενισχύσουμε τη δύναμη και τη φωνή της ενώσεως της διεθνής διαπραγματεύσεις. Και αυτό μέσω αποτελεσματικών επιδόσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα να τονίσω όλος ιδιαίτερος την ανάγκη ο πρόεδρος Μπαρόσο να αναθεωρήσει τον κώδικα συμπεριφοράς των επιτρόπων, το δελογικό κώδικα κυρίως όσον αφορά τις δηλώσεις τους για τα οικονομικά συμφέροντα τους. Ξέρουμε ότι διαπιστώθηκαν κάποια προβλήματα κατά την έγκριση από πλευρά Κοινοβουλίου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή του κ. Μπαρόσο. Της Επιτροπής Μπαρόσο. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρο, για του Ευρωπαίου συντηρητικού και μεταρρυθμιστέ. Ο κ. Τσαρνέσκι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ο Ισπανός φίλος μας, ο κ. Μένδες Δεβίγο, είπε ότι έχει πρόβλημα προσπαθώντας να εξηγήσει στην οικογένειά του τις ιδιαίτερες αυτές νομικές σχέσεις μεταξύ των διθεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Ίσως να είναι πιο υπομονετικός από μένα. Εγώ καν δεν προσπαθώ να τα συζητήσω αυτά τα θέματα με την οικογένειά μου. Είναι πάρα πολύ περίπλοκα βέβαια. Η συνθήκη της Δισαβόνα τελικά ε, είναι σαν τυφλό ραντεβού θα έλεγα. Διότι Μόλις τώρα προσπαθούμε να δούμε ποιε είναι οι αρμοδιότητε των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεω. Πολύ αργά. Καλύτερα, κάλιο αργά παρά ποτέ. Ή κάλιο αργά παρά ακόμα αργότερα. Ας μην το συζητήσουμε σαν θέμα φιλίας, α συζητήσουμε τις σχέσεις αυτές όσον αφορά πολύ ακριβείς θέσει και σχέσει μεταξύ Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συμβουλίου και Κοινοβουλίου. Καλύτερα να το συζητήσουμε έτσι πλέον επακριβώ, παρά σαν στα πλαίσια φιλία. Και τώρα για την Ευρώπη τη Δημοκρατία, ο κύριο Μέσορ Σμιτ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Σα ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε και εγώ δράτω με τις ευκαιρίες για να ευχαριστήσω τον εισηγητή για μια πολύ καλή δουλειά Είναι καλό το ότι θα παίρνουμε περισσότερη, περισσότερη πληροφορία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι πρόοδο όσον αφορά την αύξηση του κοινοβουλευτικού ελέγχου και αυτό είναι πρόοδο Και η αύξηση της διαφάνειας στη συνεργασία μας είναι και αυτό πρόοδο. Υπάρχει ένα τομέα που είναι ο σημαντικότερος από αυτού που κουβεντιάζουμε. Η κοινή εξωτερική πολιτική. Από όταν ετέθησε ισχύ η συνθήκη της Λισαβόνα, έχουμε κάποιες εξελίξεις. Εγώ την υποστηρίζω τη συνθήκη της Λισαβόνα, από τη στιγμή που δεν θα απεμπολίσουμε κυριαρχία. Ότι θα έχουμε διαβεβαιώσεις ότι κάτι τέτοιο ισχύει. Αποκτούμε μια εξουσία που δεν είχαμε πριν, την εξωτερική πολιτική. Οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί οι Ιρλανδοί είχαν πει όχι σε αυτό και προχώρησαν σε αυτή τη συνεργασία ελπίζοντας ότι η εξωτερική πολιτική θα παραμείνει στην κυριαρχία των κρατών μελών. Φαίνεται ότι τελικά αυτό θα ρυθμίζεται μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρί συμμετοχή του Συμβουλίου των ε, Υπουργών. Και αυτό είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Ο κύριο Μπρόντ έχει το λόγο τώρα για 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα αντισταθώ στον πειρασμό να απορρίψω αυτόματα σαν κάτι ανάξιο ή ύποπτο τις συμφωνίες μεταξύ δύο υποστηρικτών του προγράμματος, σχεδίου όπως αποκαλείται. Θα προσπαθήσω να δω ποιο είναι τα θετικά και αρνητικά. Η ομάδα του Κοινοβουλίου έχει αποστολή να αυξήσει τις εξουσίες του Κοινοβουλίου και την επιρροή του. Και σε κάποιο βαθμό το πετύχανε, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε. ίση αντιμετώπιση Συμβουλίου και, και Κοινοβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να εξετάζει και τι νομοθετικέ πρωτοβουλίε του ε, Κοινοβουλίου, να υπάρχουν ε, ώρε ερωτήσει με την ύπατη εκπρόσωπο και συμμετοχή σε διεθνεί διαπραγματεύσει κλπ. Υπάρχει όμω και μια άλλη όψη του νομίσματο. Η ισότητα του Κοινοβουλίου με το Συμβούλιο συνεπάγεται και μια σχετική μείωση τη εξουσία του Συμβουλίου που εκπροσωπεί έστω και άσχημα τα συμφέροντα των εθνικών κρατών η εξουσία που ασκεί το Κοινοβούλιο ασκείται δυσανάλογα από τους ηγέτες των μεγάλων πολιτικών ομάδων και των προέδρων των επιτροπών. Τα απλά μέλη αυτών των ομάδων δεν έχουν πιο μεγάλη ανεξάρτητη εξουσία από εμά που είμαστε μία εγγεγραμμένοι. Το ότι θα μπορούμε να συμμετέχουμε στις διεθνείς διαπραγματεύσεις συμπεριλαμβάνονται και συμφωνία του 2005 και το Κοινοβούλιο αντιμετωπίστηκε με περιφρόνηση. Δεν μας είπαν ποιος θα ελέγχει ε, την συμφωνία με τη ΣΥΠΑ για την ανταλλαγή πληροφοριών οικονομικού περιεχομένου. Και όταν τα μέλη τη Επιτροπή Ελευθεριών ρώτησαν γιατί υπάρχει ανάγκη απορρίτου, το μέλλον τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν απάντησε, είτε ε, γιατί δεν μπορούσε να απαντήσει, είτε γιατί υποκρινόταν ότι δεν κατάλαβε την ερώτηση. Πάμε στου άλλου αγορητέ. Πρώτο, ο κύριο Γιακολίνο έχει το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα, πώς να το πω, να συγχαρώ τους διαπραγματευτές για τα θετικά αποτελέσματα που ετέφθησαν ε, και σε σύντομα χρονικά διαστήματα. Ε, λοιπόν, η συγκεκριμένη επισφράγηση του επικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των θεσμικών οργάνων είναι αυτή η συμφωνία ε, που πιστεύουμε ότι μπορεί να εγκριθεί την Τετάρτη και να επικυρωθεί αμέσως μετά. Αυτή η συμφωνία σίγουρα δίνει όθηση στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κάτι που επιτάσσει και η συνθήκη τη Επιβάλλει μια ισχυρή συνεργασία μεταξύ των θεσμικών οργάνων και σίγουρα αυτό και προς τα εκεί κινήθηκαν οι διαπραγματευτές. Το Κοινοβούλιο δίνει, δείχνει εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα πρέπει μέσω ελέγχου συνεχούς να μπορεί να αξιολογεί τις διάφορες δραστηριότητε όσον αφορά τα εγκεκριμένα προγράμματα και τους επιτευθέντες στόχους και αποτελέσματα. Θα πρέπει να υπάρχει ιδεολογικό κώδικα για του επιτρόπου και υποχρέωση χορήγηση πληροφοριών, ακόμα και των πληροφοριών που είναι απόρριτε και εμπιστευτικέ. Εγώ δεν συμφωνώ με τι τροπολογίε που κινούνται προ αντίθετη κατεύθυνση. Οι περισσότερες όμως κινούνται προς τον κοινό στόχο. Και είμαι πεπισμένος ότι μέσω αυτού του εγγράφου θα μπορούμε να μοθετούμε καλύτερα, θα μπορούμε να αξιολογούμε και καλύτερα τον αντίκτυπο των διάφορων νομοθετικών πρωτοβουλειών. Θα ενισχυθούν οι σχέσεις με τα εθνικά κοινοβούλια ταυτόχρονα, που θα μπορέσουν να μετάχουν στις δραστηριότητες αυτές, θα μπορούν να προωθηθούν οι διάφορες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και καλύτερη διαμόρφωση πολιτικής είναι και αν αναλάβουν καλύτερα τις ευθύνες τους οι γενικές διευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εφαρμόζει από τη στιγμή που θα εγκριθεί αυτή η συμφωνία χωρίς γραφειοκρατικό τρόπο να την εφαρμόσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Γκόμα. Ένα λεπτό έχει Κυρία Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, πραγματικά η νέα συμφωνία πλαίσιο συνιστά σημαντική βελτίωση και ευάτηση των σχέσεων του Κοινοβουλίου με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε ό,τι αφορά την ειδική εταιρική σχέση βάσει τη Νική Λισαβόνα. Αυτό είναι αποτέλεσμα εξαιρετική ε, συνεργασία ε, μεταξύ Επιτροπή και τη ε, Ομάδα Εργασία του Κοινοβουλίου. Στην αναθεωρημένη αυτή συμφωνία βελτιώνεται σημαντικά η κοινοβουλευτική διαδικασία, ο κοινοβουλευτικό έλεγχο, υποχρέωση παροχή πληροφοριών και παρουσία τη Επιτροπή στον Κοινοβούλιο και καλώς ορίσατε και εσείς κύριε Επίτροπε. Θεωρώ ότι η συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις διεθνείς διαπραγματεύσεις είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα προς τα εμπρός που θα διευκολύνει τον, ε, διευκολύνει το στόχο ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να έχει μεγαλύτερη συμμετοχή στις διαδικασίες. Ε, θα πρέπει να δούμε επίσης και την συνέχεια, πώς θα ενημερώνετε για τη συνέχεια που δίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις διάφορες υποθέσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να μας κάνει μετά από ένα χρόνο μία πρόταση νομοθετική και να παρουσιάσει τα επόμενα προγράμματα εργασίας. Και αν δεν κάνει πρόταση θα πρέπει να εξηγήσει αναλυτικώς τους λόγους στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ελπίζω επίσης ε, να αντιμετωπιστεί με τον θέοντα σεβασμό ε, και το θέμα των πρωτοβουλίων των Ευρωπαίων ε, πολιτών. Εγώ πραγματικά ε, θεωρώ ότι η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα ακολουθήσει, θα εγκρίνει τα αποτελέσματα των διαπραγματεύσεων Επιτροπής και Ομάδας Εργασίας του Κοινοβουλίου. Ο κύριος Κόλμαν, ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε. η συμφωνία για τη σχέση μεταξύ της Κομισιόν και του Σώματος όσον αφορά την ε, συνθήκη της Λισαβόνας και υποτίθεται ότι αυτό θα οδηγήσει σε πιο δημοκρατική διαδικασία. Αυτό όμως είναι μια ουτοπία δημοκρατίας που δεν υπάρχει. Και θα σας πω γιατί. Η Λισαβόνα δεν έχει δημοκρατική ηθική ισχύ στο Ηνωμένο Βασίλειο όπου οι απλοί πολίτες έχουν εξαπατηθεί από την κυβέρνηση και δεν μπορούσαν να πούνε την άποψή τους. στην πράξη θα συγγενήσουν τα πράγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως είχαν στα παρασκήνια και κλεισμένων των θερών κλπ. Εν ευθέτω χρόνο ε, θα καταψηφίσουμε εμείς αυτές τις προτάσεις μια που δεν αναγνωρίζουμε τη Λισαβόνα εκτός εάν υποβληθεί στον ε, λαό του, της Βρετανίας για να ακούσουμε τη δική τους άποψη. Αυτή είναι η δημοκρατία. Ευχαριστώ, λέει πρόεδρος, η κυρία Φρασικό Φαβένοβα για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Χαίρομαι ιδιαίτερα που σήμερα μπορούμε να συζητήσουμε την αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτή η αναθεώρηση επιβεβαιώνει και διευκρινίζει την ισχυρότερη θέση του Κοινοβουλίου μετά τη συνθήκη τη Λισαβόνα. Θα ήθελα ειδικότερα να τονίσω τη συμφωνία μεταξύ τη Επιτροπή και της Ομάδας Εργασίας ε, του Κοινοβουλίου για τη συμφωνία πλαίσιο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Αντιπρόεδρο τη Επιτροπή για την συμμετοχή του στι εργασίε αυτέ. Δύο λόγια τώρα για τη συμφωνία πλαίσιο. Ισχυρότερη θέση του Κοινοβουλίου κάνει πιο δημοκρατική την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμεί που έχουμε εκλεγεί από του πολίτε των κρατομιλών της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμμετέχουμε στη βελτίωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ε, και θα έχουμε ε, λόγο, ε, θα είναι υπόλογη η Επιτροπή απέναντί μας σε ό,τι αφορά τα ειδικά μέτρα το οποίο θετεί σε σχέση με οποιοδήποτε νομοθετικό αίτημα. Ταυτόχρονα θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ζητά και το πράσινο φως για αλλαγή του κώδικα διοντολογίας. Θεωρούμε ότι στο πλαίσιο αυτής της συμφωνίας πλαίσιο θα ενημερώνεται καλύτερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και για εκκρεμής διαπραγμάτευση διεθνείς συνθήκες. Υπάρχουν αρκετά μέτρα στο πλαίσιο της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου και είμαι πεπισμένη ότι όλα αυτά θα έχουν ως αποτέλεσμα την πιο αποτελεσματική και στενή συνεργασία των δύο θεσμικών οργάνων και θα οδηγήσουν σε μια συνεκτική εφαρμογή της συνθήκης της Λισαβόνας. Τέλος, ήθελα να τονίσω έναν άλλο σημαντικό τομέα ένα μέτρο πολύ σημαντικό που θα ε, εξασφαλίσει την συνεργασία με των πολιτών, που θα είναι η εφαρμογή των πρωτοβουλειών των Ευρωπαίων πολιτών. Κύριε Σόβατα, ευχαριστώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την ε, έκθεσή του και τον κύριο ε, Σεφκοβίτσι για τις διαπραγματεύσεις που είχαμε. Δεν ήταν εύκολος, αλλά δίκαιος διαπραγματευτής. Και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα είναι βέβαια η βάση της συνεργασίας μας και η ερμηνεία που δίνει ο κύριος Ράντζελ είναι κάπως αναλυτική, αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποιους ε, στόχους μπροστά μας. Αυτό που παραμένει ε, είναι ότι ε, δεν πρέπει να έχουμε μόνο διαφάνεια μεταξύ μας, αλλά και με το Συμβούλιο που απουσιάζει ότι αν εμείς συνεργαζόμαστε ε, καλά θα μπορέσει και το Συμβούλιο να συνεργαστεί. Το Συμβούλιο δεν είναι εντύπωση σαν παιδί που του πήραν το παιχνίδι και κλαίει τώρα και διαμαρτύρεται. Αντί να κάθε να κλαίει θα πρέπει να καταλάβει ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι το καλύτερο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Αν θέλουμε να είμαστε ισχυροί προς τα έξω, εάν θέλουμε η κοινή εξωτερική πολιτική να είναι σημαντική και κοινέ συμφωνίε εξωτερικού εμπορίου, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την καλή συνεργασία μαζί μας. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Ο κύριο Σαρίφ, ένα λεπτό. Κυρία Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ξέρουμε όλη τη συνθήκη τη ε, της ενισχύει τι εξουσίε του Κοινοβουλίου. Λίγοι από εμά έχουμε επίγνωση για τι ριζικέ αλλαγέ που επιφέρει, κυρίω όσον αφορά τον τομέα τη εμπορική πολιτική που παρακολουθώ η συνθήκη της Λισαβόνας θα, θα, θα επικοινώνει ό,τι μπορικές συμφωνίες της διεθνής λόγω της συμφωνίας αυτές. Έχουμε τη συμφωνία με την Κορέα της Ελευθέρων Συναλλαγών και είναι το πρώτο μήνυμα δημιουργία να ταραχεί. Αλλά οι σοσιαλιστές και δημοκράτες θέλουν να προχωρήσουν περισσότερο από αυτό που προβλέπει η συνθήκη. Εγώ με το φερέφωνό τους και παρά τον σκεπτικισμό κάποιων που έχουν αντιρρήσει και άλλων που έχουν αντιρρήσει, εγώ στέλνω σαφέ μήνυμα. Το Κοινοβούλιο πρέπει να επικυρώσει κάθε εμπορική συμφωνία, θα πρέπει να συμμετέχει από την αρχή τη διαδικασία. διαδικασία. Αυτό που θα πρέπει. Αλλιώ θα είναι τοπικέ οι σχέσει με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Διότι θα πρέπει να ε, ενημερωνόμαστε πλήρω. Και καλό και το Συμβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουν να σέβονται το πνεύμα το κοινοτικό και το δημοκρατικό, τη δημοκρατική πνοή των συνθήκων. Ε, διότι έχουμε ένα σύνδρομο τη Στοκόλμη όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο. Οπότε προσέχουμε. Θα πρέπει να χρησιμοποιούμε όλα τα δικαιώματά μα, διότι είναι και δικαιώματα των πολιτών μα. Σα ευχαριστώ. Ο κύριο Μιλάνα, ένα λεπτό. Ναι. Η αναθεώρηση αυτή τη συμφωνία μεταξύ Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέτει τι βάσει για καλύτερη συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων. Πάρα πολλέ προόδοι επετέφθησαν για τη διαδικασία, για τον αθωματικό σχεδιασμό, για τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, για τι υποχρεώσει ε, χορηγή πληροφοριών. Η παρουσία τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Κοινοβούλιο καλύπτεται. Αλλά αυτό που θεωρώ ότι πρέπει να υπογραμμιστεί περισσότερο αναφέρεται στι προόδου που πετέχθησαν στον τομέα τη διοργανική διαστάσεω όσον αφορά τι διεθνεί σχέσει ο ρόλος που ανατίθεται στο Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να θεωρηθεί κάτι που ενισχύεται. Είναι κάτι που ήταν υποχρέωση. Κανεί δεν πρέπει να αμφισβητεί ότι θα πρέπει να υπάρχουν παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στι διάφορε διεθνεί διασκέψεις, στις πολυτερεί και τι διμερείς και ότι είναι μια πράξη ευθύνη αυτή. Το να ανηθούμε το καθεστώ των παρατηρητού των βουλευτών στι συζητήσει για διμερείς συμφωνίε, όπω είναι οι ελευθερικέ συμφωνίε, στερεί εκ των πραγμάτων μια επίγνωση των γεγονότων τη διαπραγματεύση, που θα πρέπει μετά να τοποθετηθεί το Κοινοβούλιο σε αυτέ τι συμφωνίε. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα λιγότερο από αυτά που βλέπετε, διαφορετικά θα πρέπει απλώ να επικυρώνουμε διμερεί συμφωνίε σε κοινοβούλιο, που δεν μπορούν να τροποποιηθούν. Θα πρέπει να μπορούμε να συμμετέχουμε στι διαπραγματεύσει. Και να μην είναι απλώ τυπική επικύρωση μετά ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Περνάμε στη δικασία Κατσιάη. Η κυρία Ρόιτοβα έχει πρώτο λόγο για ένα λεπτό. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι καλό που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταλαβαίνει ότι για να έχουμε επιτυχία στο μέλλον θα πρέπει οι αποφάσει να λαμβάνουν κατά δυνατόν την τρόπο. Θα πρέπει δηλαδή να ενδυματωθεί ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η νέα συμφωνία με την Κομισιόν ε, ενισχύει τη θέση του Κοινοβουλίου πέρα από αυτό που προβλέπει η συνθήκη της Λισαβόνας. Χαίρομαι που θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερες εκθέσεις ε, ε, επιπτώσεων, θα υπάρχουν περισσότερες αποφάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα πρέπει οι βουλευτές πραγματικά να έχουν στα χέρια τους μεγαλύτερη ελευθερία στην μελέτη των εγγράφων. Δεν θα πρέπει να επικαιρώνουν τυπικά, θα πρέπει να έχουμε πραγματικά όλες τις πληροφορίες στα χέρια μας για να μπορέσουμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων να επιδράσουμε στις αποφάσεις. Στο μέλλον, η Κομισιόν και το, Κοινοβούλιο, και το Συμβούλιο θα πρέπει να συνεδριάζονται πολύ καλύτερα με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ, Λίπρο. Και θα πάρει κανένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η συνθήκη της Λισαβόνας ε, έχει πλέον ε, ορίσει νέες ευθύνες και υποχρεώσεις και για το Κοινοβούλιο και για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και είναι πολύ καλό το ότι μετά από ένα χρόνο από την θέση σε ισχύ της συνθήκης θα έχουμε αναθεώρηση τη Συμφωνίας Πλαισίου ώστε να μπορέσουμε να εκπληρώσουμε καλύτερα τους, ε, τα κοινά μας καθήκοντα. Η Συμφωνία για Κοινέ Διαδικασίες θα καταστήσει δυνατή την αποτροπή παρεξηγήσεων κατά τη λήψη αποφάσεων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται σε συμφωνίε μεταξύ κρατών. Κάποιε από τι αρμοδιότητε έχουν χωρίσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο ε, Κοινοβούλιο τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό λοιπόν η συνθήκη τη Λισαβόνα ε, συνεπάγεται κάποιε ευθύνε και ό,τι αφορά τη συνεργασία με τα εθνικά κοινοβούλια. Θα πρέπει λοιπόν για τη σωστή συνεργασία να καθορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται αυτή και θα πρέπει να το λάβει υπόψη και η Επιτροπή. Ευχαριστώ, ο Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συνεργάζονται ε, και υποτίθεται ότι είναι δημοκρατικά βασισμένοι. Η Κομισιόν όμως που δεν έχει δημοκρατική βάση είναι το όργανο που υποβάλλει τις προτάσεις για τους νόμους, κανονισμούς και οδηγίες του της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν ελλείψεις ε, στη συνθήκη της Λισαβόνας. Για να μπορέσει σωστά να εργαστεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να έχει και τη δυνατότητα να έχει περισσότερες πληροφορίες. Σύμφωνα με την νέα διαδικασία θα πρέπει πρόσωπος του λαού, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δηλαδή, να εμπλέκεται στη διαδικασία των νωρίτερων δυνατών. Και έτσι θα πρέπει να ενδυναμωθεί το Κοινοβούλιο και θα πρέπει η η εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής να μην παραμένει στα χέρια της υπηρεσία εξωτερικής δράσης μόνο. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Μπαζέσκου, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ. Θεωρώ ότι η νέα συμφωνία θα βελτιώσει σημαντικά τις σχέσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο 2010-2015. Η αναθεώρηση της νομικής βάσεως όσον αφορά τη συνεργασία αυτή φτάνει την κατάλληλη στιγμή. Λίγο χρόνο μετά τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της ε, Λισαβόνας. Οι νέοι κανόνες καθορίζουν σαφώς τις πολιτικές ευθύνες των δύο θεσμικών οργάνων και ενισχύουν τις αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αρμοδιότητε που απέκτησε πρόσφατα όσον αφορά τι διαδικασίε λήψη αποφάσεω. Λόγω τη ισότιμη αντιμετωπίσεω, το Κοινοβούλιο θα έχει τα ίδια δικαιώματα όπω και το Συμβούλιο όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα ε, για τα θέματα τα νομοθετικά και του... τα δημοσιονομικά και θα μπορεί να συμβάλλει στη διαμόρφωση των προγραμμάτων των ετησίων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, ενισχύοντας τη συμμετοχή των πολιτών στη διαμόρφωση προτεραιοτήτων των πολιτικών των Ευρωπαϊκών. Ευχαριστώ. Τελευταία στη διαδικασία Κατσουδιά, κυρία Μομπάη, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όσον αφορά το θέμα που συζητούμε, πρέπει να πω Λέμε ότι ένα κακό, ξέρουμε ότι ένα κακό δέντρο κάνει έναν κακό καρπό, καλό δέντρο κάνει καλό καρπό. Λοιπόν, ε, θα έπρεπε να ακολουθήσουμε σωστή προσέγγιση έχουν στα αποτελέσματα. Ε, είχαμε, κατά το, υποχρεωθήκαν τα κράτη-μέλη με δικτατορικό τρόπο να υπογράψουν τη συνθήκη της Λισαβόνας παρά τη βούληση των πολιτών, τουλάχιστον όσον αφορά τη χώρα μου, την Ουγγαρία. Πάρα πολλά θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών ε, ε, απομακρύθηκαν τα κράτη-μέλη και πήγαν στις Βρυξέλλες. Όσον αφορά το δίκαιο συνθήκη της Λισαβόνας δεν ισχύει στην Ουγγαρία όσον αφορά το δίκαιο της χώρας μας διότι δεν ελήφθησαν οι υπόψη οι απόψει των πολιτών δεν έγινε καμία διαβούλευση με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις και μεταξύ άλλων εάν ψηφίστηκε αυτή η συνθήκη χωρίς να γνωρίζει κανείς το περιεχόμενο του κειμένου. Αυτές είναι συνέπειες μια συνθήκη που πέρασε δικτατορικά. Και ο Τιο Εύκοβιτς, ο κόσμος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους ομιλητές, κυρίως που που υποστήριξαν την συμφωνία πλαίσιο, ε, διότι πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το πλαίσιο για να μπορέσουμε να συνεργαστούμε καλύτερα στο μέλλον. Θα ήθελα εκ νέου να υπογραμμίσω τις, ε, την ευγνωμοσύνη μου προς την ομάδα εργασίας, την ομάδα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Περάσαμε πολύ χρόνο μαζί. Ε, περάσαμε ώρες εντατικών διαπραγματεύσεων. Νομίζω ότι αυτή η δουλειά απέδωσε και σήμερα μπορούμε πράγματι να χαιρετήσουμε μια έξοχη συμφωνία. Άκουσα με τα μεγίστη προσοχή στα σχόλια των αξιοτήμων μελών και τι ερωτήσει που ακούστηκαν που αντικατοπτρίζουν κάποιε ανησυχίε για την σα συμφωνία. Και γι' αυτό θα ήθελα καταρχά να υπογραμμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι αυτή η αρχή που θεσπίζεται είναι πολύ σημαντική. Δηλαδή, για τη συνεργασία μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων, το η αναθεωρημένη συμφωνία πλαίσιο δεν θα πρέπει να μας απομακρύνει από τα επιτευθέντα θετικά αποτελέσματα. Εφαρμόζοντας τη συμφωνία πλαίσιο, σε όλες τις περιπτώσεις θα καταλήγουμε σε σαφείς βελτιώσεις. Το τούτων λεχθέντων και τα δύο μέρη παραδέχτηκαν για τι διαπραγματεύσει ότι αντιμετωπιστούν δυσκολίε όσον αφορά την ερμηνεία τη συμφωνία, αλλά εξέφρασαν την προθυμία να εφαρμόσουν την αναθερημένη συμφωνία πλαίσιο με τον πλέον επικοδομητικό τρόπο. Και σα διαβεβαιώνω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δεσμευμένη να το κάνει αυτό. Αξιότιμα μέλη, Είμαι πεπισμένο ότι στην πράξη θα δούμε ότι πολλές ανησυχίε που εξεφράσαν σήμερα δεν θα αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Αλλά ε, θα πρέπει να προχωρήσουμε και πιο πέρα από τις ευθύνε που δίνουν οι συνθήκε στα διάφορα ε, θεσμικά όργανα και ανισορροπίες θα πρέπει να αποκατασταθούν. Ακούστηκαν διάφορε ανησυχίε όσον αφορά τη δήλωσή μου ότι το διευθυντικό κώδικα, το υποστηρίξατε αυτό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πράγματι σύντομα θα υποβάλει σχετική πρόταση για ε, αναθεωρημένη αναθεώρηση του δεντολογικού κώδικα και σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πλαίσιο θα ζητήσει και την γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έγκαιρα. Κάτι που υποσχεθήκαμε άλλωστε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων. Κλείνοντα λοιπόν, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω το εξή. Εάν ανακαλύψουμε τυχόν προβλήματα, ξανά θα καθίσουμε όλοι μαζί για να βρούμε κάποια λύση. Και μάλιστα προβλέψαμε αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου ήδη μέχρι το τέλος του 2011. Άρα θα έχουμε δυνατότητες να διορθώσουμε τυχόν λάθη. Και εν αυτή τη ενία προσβλέπω σε συνεργασία μαζί σας επί τη βάση της αναθεωρημένης συμφωνίας πλαισίου και περιμένω ότι θα υποστηρίξετε αυτή τη συμφωνία τελικά την Τετάρτη. Πιστεύω και ελπίζω ότι αυτό το θετικό πνεύμα θα επικρατήσει και στις γενικότερες σχέσεις μεταξύ όλων των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, διότι αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμά και αυτό θα πρέπει τελικά να πετύχουν. Ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Τώρα ο συγχητής έχει πάλι το λόγο. Παρακαλώ κύριε Ρέντζελ. Ε, δύο λεπτά. Ε, σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στα όσα άκουσα κατά τη διάρκεια της συζήτησης και θέλω κυρίως να ε, τονίσω το εξή. Ένα στόχος του συμφωνίας αυτής πλαίσιο ήταν ε, σε θέμα κοινή νομοθεσία και ε, θέματα προπολογισμού να τεθούν επίσης ώρες ε, το Κοινοβούλιο και η Επιτροπή. Για τα άλλα θέματα θελήσαμε επίσης να σεβαστούμε την ισορροπία αρμοδιοτήτων που προβλέπεται από τη δίκτυες της Λισαβόνας σεβόμενη την αρχή της ε, ε, κατανομής των αρμοδιοτήτων ούτως ώστε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μπορεί καλύτερα να ασκεί τον πολιτικό του έλεγχο. Νομίζω ότι αυτή η διευκρίνηση, αυτές οι εξηγήσει δηλαδή που δίνει το η αναθερημένη συμφωνία πλαίσιο, είναι θετικές. Αυτή η εξέλιξη είναι πολύ καλή για τα θεσμικά όργανα. Οι σχέσει του είναι πιο σαφείς και πιο διαφανείς. Αυτό είναι καλό μας και για τα άλλα θεσμικά όργανα, συγκεκριμένα δηλαδή για το Συμβούλιο. Γιατί τώρα πια το Συμβούλιο έχει στη διάθεσή του μία καθαρή εικόνα του τρόπου με τον οποίο θα διαμορφωθούν οι σχέσεις Κοινοβουλίου και Επιτροπής μετά τη θέση ισχύ της συνθήκης του Λισαβόνας. Γι' αυτό, εάν ίσως πολλές φορές ίσως το Συμβούλιο εξέφρασε κριτική κατά του αναθεωρημένου ε, σχεδίου πλαίσιου, εγώ πιστεύω ότι τα αποτελέσματα είναι θετικά για όλα τα θεσμικά όργανα και θα έρθει εκείνη η μέρα κατά την οποία θα δούμε ότι το αναθεωρημένο σύμφωνο πλαίσιο είναι όχι μόνο προς όφελος των πολιτών, αλλά προς όφελος και των τριών θεσμικών οργάνων της Ένωσης, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα της συνθήκης της Λαβώνας. Και ευχαριστώ την Κομισιόν για το πνεύμα συνεργασίας που έδειξε. Ευχαριστώ όλοι οι πρόεδρος. Ολοκληρώνεται η συζήτηση. Ψηφοφορία θα γίνει στις, την Τετάρτη στις 12 το μεσημέρι. Λοιπόν, αξιότιμοι συνάδελφοι, περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης.